Μπορούμε να ξεκινήσουμε τις ε, απομοκευματινές μας ε, συνεργασίες, την απογευματινή μας συνεδρία. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την παρουσίαση από τον κύριο Καμάλ Χωσέιν, πρόεδρο της ε, Euromet, μια παρουσίαση λέω σχετικά με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Μετρολογίας για την καινοτομία και την έρευνα. Θα δώσουμε αμέσως το λόγο για 20 λεπτά στον κύριο Χωσέιν. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα σε όλους σας. Πρώτα απ' όλα, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Θεωρούμε ότι είναι μεγάλη τιμή να έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για εσά, για, εμνόπιόν σας για αυτά τα νέα ε, προγράμματα. Έχω μαζί μου τον κύριο Στέγκερ, ο οποίος είναι πρόεδρος του ε, EMPIR και τον ε, καθηγητή Γιάνκο Πρόστσεκ. Θα πάρουν τον λόγο μετά. Δεν, θα σας δυσκολέψω πάρα πολύ ε, μιλώντας για τη μετρολογία, γιατί είναι από τα θέματα που μπορεί να αποθαρρύνουν ε, τον κόσμο. Ε, γιατί στην, λοιπόν, η μετρολογία ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι ασχολείται με τον καιρό, αλλά ούτως ή άλλως σήμερα δεν το χρειαζόμαστε, είναι πολύ καλός ο καιρός, δεν έχουμε πρόβλημα. Η μετρολογία λοιπόν αφορά τις ε, μετρήσεις. Είναι ε, αυτά, ένα από αυτά τα στοιχεία τα οποία δεν γνωρίζει ο κόσμος ε, και στο Ηνωμένο Βασίλειο λέμε ότι είναι ο αφανής σύρος η μετρολογία, είναι αυτός που κάνει τα πάντα αλλά ο κόσμος δεν ξέρει ότι, είναι, ότι υπάρχει και ότι κάτι κάνει και ότι βοηθάει την κοινότητα. Έχω εδώ διάφορα slides, ε, διάφορες διαφάνειες, ε, οι οποίες αναφέρουν ε, παραδείγματα. Λοιπόν, όταν βάζετε πούμε, βενζίνη στο αυτοκίνητό σας, βάσει της μετρολογίας έχετε τη διασφάλιση ότι πληρώνετε ακριβώς για το ποσό το οποίο έχετε για το για τον όγκο που έχετε ε, βάλει. Εάν κάποιος ατυχώς έχει καρκίνο, ε, τότε ε, βάσει της μετρολογίας μπορεί να οριστεί τι θεραπεία θα πάρει, σε ποιο βαθμό, έτσι ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί ο όγκος, αλλά να μην πάθουν τίποτα τα υγιή κύτταρα και τέλος πάντων να μην έχει πρόβλημα ο ασθενής. Επίσης, θα δείτε ότι πολλή συζήτηση ε, γίνεται ε, για την ε, για το κλίμα, για την αλλαγή της ε, θερμοκρασίας, αν ανεβαίνει. Ε, ενδεχομένως, ε, εάν περιμένουμε να αυξηθεί η θερμοκρασία για να καταλάβουμε τι γίνεται, τότε το Λονδίνο και το δικό μου το σπίτι θα βρεθεί κάτω από το νερό. Θα έχει πλημμυρίσει το Λονδίνο μέχρι να καταλάβουμε τι γίνεται. Άρα πρέπει εκ των προτέρων να κάνουμε τις μετρήσεις. Επίσης, βασική επιστήμη. Ε, ας πούμε την... Ε, about the news headline that came... τις σταθερές μεταβλητές της φύσης. Πριν από μερικούς μήνες ε, ε, ίσως έξι μήνες πριν και πάνω, ε, έγινε λόγος για ένα πείραμα ε, στην, στη Γενέβη και για να μετρηθεί το, ότι, το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν ότι τα πράγματα μπορεί να ταξιδεύουν πιο γρήγορα με μεγαλύτερη ταχύτητα από το φως έπρεπε να γίνουν σωστές μετρήσεις. Πρέπει λοιπόν σε κάθε περίπτωση να έχει κανείς καλές μετρήσεις. Όταν έχει κανείς ας πούμε τα φωτοβολταϊκά στο, τα πανέλα αυτά ε, στην οροφή του σπιτιού του και εκεί πρέπει να ξέρει ότι λειτουργούν σωστά στις μεταφορές, ε, τα οχήματα, τα αεροπλάνα. παλιότερα για να μπορούν να λειτουργούν καλά θα έπρεπε να έχουν γίνει ε, πάρα πολλές ε, μετρήσεις. Τώρα μπορούμε με πολύ εύκολο τρόπο να κάνουμε όλες τις μετρήσεις που χρειάζονται έτσι ώστε να λειτουργούν τα πράγματα σωστά. Κάτι άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι η ζήτηση για σωστές μετρήσεις αυξάνει. Από τη μία πλευρά λοιπόν έχουμε την τεχνολογική όθηση ε, η οποία απαιτεί όλο και περισσότερο ε, εξειδητημένες μετρήσεις αλλά χρειάζεται και μεγαλύτερη γνώση έτσι ώστε να κατανοήσουμε ε, τι είναι αυτές οι συνθήκες, ποιες είναι οι μετρήσεις και ποιες είναι οι απαιτήσει των μετρήσεων. Ε, σε όλο το φάσμα της ζωής μας, ε, όλο και περισσότερο χρειαζόμαστε μετρήσεις, ε, σωστές, ακριβείς, καλύτερες μετρήσεις. Μερικές φορές ο κόσμος ταυτίζει τη μετρολογία με τα πρότυπα και θεωρεί ότι δεν είναι και τίποτα τρομερό. Αλλά παρασάγκας απέχει. Ε, θα δείτε ότι έχω εδώ ένα γράφημα το οποίο στο οποίο αναφέρεται ότι, το οποίο αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο από την ε, ιδέα πηγαίνει κανείς στην πραγματοποίηση γιατί όλοι πιστεύουν οι περισσότεροι ότι η καινοτομία προέρχεται από την ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά ε, σκεφτείτε ας πούμε τα ηλεκτρονικά ε, χρειάζεται κάποιος να τα κάνει και πριν ξεκινήσει ο έλεγχος, το σύστημα παραγωγής τώρα ειδικά που τα πράγματα έχουν όλο και μικρότερο όγκο, κάποιος πρέπει να κάνει τις σωστές μετρήσεις. Ολόκληρη η αλυσίδα λοιπόν από την σύλληψη της ιδέας μέχρι ε, το αντικείμενο που θα βγει στην πραγματική ζωή και θα κυκλοφορήσει χρειάζεται τη μετρολογία και οι καμπύλες δείχνουν ότι βεβαίως στο αρχικό στάδιο της σύλληψης είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά στην άλλη πλευρά ε, της ε, αλυσίδας, ε, όσον αφορά την ετοιμότητα δηλαδή της τεχνολογίας, εκεί παίζει μεγάλο ρόλο η μετρολογία και άλλωστε αυτό και η Νέστα στον Ηνωμένο Βασίλειο πρόσφατα το αναγνώρισε. Όσον αφορά λοιπόν την μετρολογία έχουμε τώρα ένα πρόγραμμα το οποίο είναι το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Μετρολογίας. Θα πω δύο λόγια για αυτό το νέο πρόγραμμα. Έχουμε 30 ε, προγράμματα τα οποία λειτουργούν ήδη στα πλαίσια του, Ευρωπαϊκού του νέου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Μετρολογίας για την καινοτομία και την έρευνα και έχουμε μερικά πολύ καλά παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο ε, συγκεκριμένα η Μητρολογία βοηθάει την υλοποίηση νέων καινοτόμων ε, συγγνώμη, προϊόντων τα οποία έχουν σχεδιαστεί αλλά πρέπει να φτάσουν στην αλυσίδα παραγωγής. Αυτά όσον αφορά την καινοτομία. Εδώ έχω ένα σχεδιάγραμμα Αν δείτε λοιπόν αυτό το σχεδιάγραμμα, ε, στο, στην κορυφή αναφέρονται οι μεγάλες προκλήσεις ε, της πολιτικής και της ε, κοινωνίας ε, δηλαδή όλα, όλα αυτά τα στοιχεία για τα οποία θέλουν συγκεκριμένες ε, ρυθμίσεις και δεσμεύσεις. Ας πούμε λέμε ότι ε, δεν πρέπει να υπάρχει εκπομπή συγκεκριμένης ουσίας παραπάνω από τόσο στη δεξιά πλευρά του γραφήματος ε, βλέπετε ότι αναφέρω τη λέξη ε, κανονισμός. Είναι η ρύθμιση λοιπόν η οποία μπορεί να γίνει μέσω των κανόνων, των ορίων ασφαλείας, ε, όλων αυτών των εξειδικεύσεων που θα πρέπει μέσα από διαφάνεια και μετά τις προτύπων να αναφέρεται. Αλλά τα πρότυπα πώς μπορούν να εφαρμοστούν μόνο μέσα από σωστή και αξιόπιστη μέτρηση. Έτσι λοιπόν το ένα κομμάτι του παζλ έρχεται και δένει με το άλλο. Ε, δηλαδή οι ίδιες, η ίδια η κοινωνία μέσω των προσπαθειών που κάνει για να φτάσει σε, στην αντιμετώπιση κάποιων προκλήσεων χρειάζεται να αναπτύξει και άλλα ε, ε, στοιχεία, την τυποποίηση, την πιστοποίηση, την μετρολογία. Η τυποποίηση πάντως δεν είναι, ε, ε, ε, η μετρολογία δεν μπορεί να κατεβεί μονάχα στο επίπεδο της, του ορισμού προτύπων, είναι κάτι πολύ περισσότερο. οι οργανώσει τώρα, οι οργανισμοί που ασχολούνται με τη μετρολογία. Εμείς είμαστε το Euromet. Θα πω δύο λόγια για το Euromet μετά. Ε, τα μετρολογικά Ινστιτούτα ε, είναι ε, καταναμημένα σε διάφορες περιφέρειες, στις Ηνωμένες Πολιτείες, Νότια Αμερική, Αφρική κτλ. Η EuroMet είναι λοιπόν μία τέτοια περιφερειακή οργάνωση. Τα Εθνικά Ινστιτούτα Μετρολογίας της Ευρώπης έχουν αρχίσει να δουλεύουν, να συνεργάζονται μεταξύ τους από το 1900 σχεδόν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 και το Euromet ξεκίνησε ήδη από το 1999 ή κάπου εκεί και έγινε Euromed όπως είναι τώρα δηλαδή το 2007. Ε, οι 23 χώρες ε, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν συμφωνήσει να συμμετάσχουν και συμμετέχουν στο νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Μετρολογίας για την Καινοτομία και την Έρευνα. Έχουμε και πέντε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή, Ένωση, συγγνώμη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί. Ε, τα προγράμματα αυτά. Ε, η Κομισιόν μάλιστα έδωσε ε, την χρηματοδότηση στην Euramet η οποία διαχειρίζεται το προϋπολογισμό μόνη της και η Euramet έπρεπε να δημιουργήσει μια οντότητα η οποία να μπορεί να είναι σε θέση να λειτουργήσει τον προϋπολογισμό αυτό. Λοιπόν, Είπαμε ότι 23 ε, χώρες ε, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την καινοτομία και την έρευνα. Συνεργαζόμαστε επίσης με Ινστιτούτα τα οποία δεν είναι εθνικά Ινστιτούτα Μετρολογίας απαραίτητα, αλλά είναι σε μερικές περιοχές πάρα πολύ σημαντικά. Η συνεργασία σε θέματα μετρολογίας είναι πάρα πολύ σημαντική και για την Ευρώπη. Έχω και μια διαφάνεια που ενδεχομένως θα σας δώσει καλύτερα να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Πάντως ξεκινήσαμε ε, μια συνεργασία το 2002 και περάσαμε από διάφορα στάδια ευρωπαϊκής ε, συνεργασίας. Το 2002 είχαμε το πρόγραμμα ε, ΙΡΑ μέρα μάλλον. Μετά είχαμε το Αϊμύρα με περισσότερους, μετά είχαμε μεγαλύτερη συνεργασία, το λεγόμενο πρόγραμμα Αϊμύρα Plus, μετά είχαμε το EMRP ε, για την περίοδο 2009-2013 ακόμα περισσότερα ε, μέλη και τώρα στο EMPIR e ακόμα περισσότερες ε, χώρες και μεγαλύτερο προπολογισμό. Σιγά σιγά δηλαδή ενθαρρύνθηκαν και άλλες χώρες να συμμετάσχουν. Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα έχουμε 28 από τις 28 χώρες μέλη που θα θέλουν να συνεργαστούν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι σημαντικό και για την, ευρωπαϊκή, την αγωνιστική πραγματικότητα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργείται ένα κατάλληλο περιβάλλον ε, βάσει της ανάπτυξης μετρολογίας έτσι ώστε ο ανταγωνισμός ε, με τις ΗΠΑ ας πούμε ή άλλες περιοχές του κόσμου να είναι σωστή. Ε, έχουμε 28 χώρες που συμμετέχουν λοιπόν, που θα συμμετάσχουν στο ε, EMPIR και ελπίζω ότι θα αυξηθεί ο αριθμός. Λοιπόν, το πρώτο πρόγραμμα, αυτό το Aimira Plus, ε, ολοκλήρωσε 21 projects με χρηματοδότηση 63 εκατομμυρίων. Τώρα έχουμε ξεκινήσει για το τελευταίο μας πρόγραμμα τη διαδικασία επιλογής. Όσον αφορά τώρα τις εξωτερικές συνεργασίες, έχουμε 128 μεγάλες εταιρείε ε, οι οποίες ε, συνεργάζονται, 125 μάλλον. Έχουμε μικρομεσαίες εταιρείε 62, ε, έχουμε 123 ε, συνεργάτες οι οποίοι έχουν υπογράψει ήδη συμβάσεις ε, ότι δηλαδή θα ε, παραδώσουν το, την εργασία τους χωρίς να έχουν άμεση χρηματοδότηση. Αυτό, είναι, αυτό δείχνει μάλλον και πόσο σημαντικό είναι το πρόγραμμα. Δηλαδή συμμετέχουν ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι δεν θα έχουν καμία χρηματική απολαβή από το πρόγραμμα αυτό. Αλλά παρόλα αυτά δεσμεύονται ότι θα κάνουν τη δουλειά τους θα την παραδώσουν έγκαιρα. Έχουμε ε, περίπου 900, ε, χίλιους μάλλον ε, εμπλεκόμενους φορείς οι οποίοι είναι ήδη ενεργοί. Και πρέπει να πω ότι είμαι βέβαιος ότι θα αυξηθεί, θα διπλασιαστεί ο αριθμός αυτός. Βεβαίω τα πανεπιστήμια είναι πάρα πολύ σημαντικά, από εκεί ξεκινάει η νέα γνώση, από εκεί ξεκινούν τα προγράμματα που θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω. Και πρέπει να πω ότι κάθε χώρα έχει το δικό της Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας ε, που είναι υπεύθυνο. Όταν λέμε τι ώρα είναι, ε, η κάθε χώρα έχει τα δικά της πρότυπα για την ώρα και συντονίζονται όλοι αυτοί μεταξύ τους έτσι ώστε να ξέρουμε ότι η ώρα είναι η σωστή. Ε, γιατί φανταστείτε, ξεκινά ένα ταξίδι αεροπορικό από τι Βρυξέλλε στο Λονδίνο, θα ήταν πάρα πολύ δυσάρεστο ε, τα ρολόγια να μην ταυτίζονται. Αυτό συμβαίνει γιατί τα Εθνικά Ινστιτούτα Μετρολογία συνεργάζονται. Ε, απ' την άλλη πλευρά όμως είπαμε νέα γνώση ξεκινάει από τα πανεπιστήμια ε, και εμείς με τη δικιά του συμβολή, με το δικό τους ε, input έχουμε την δυνατότητα να βοηθήσουμε έτσι ώστε, όλοι, έτσι ώστε το επίπεδο της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης να είναι σημαντικό. Αυτό είναι το output, το αποτέλεσμα που έχουμε. Όσον αφορά το νέο πρόγραμμα, Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει συμφωνία και ελπίζω και ότι η Επιτροπή θα το στηρίξει. Αν μπορείτε με οποιοδήποτε τρόπο να μας βοηθήσετε θα το εκτιμήσουμε ιδιαίτερος. Ε, πρέπει να υλοποιηθεί το πρόγραμμα αυτό σαν πρωτοβουλία του άρθρου 185. Ε, μιλάμε για ένα συνολικό ε, ποσό 600 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ των χωρών Euramet και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι εδώ ε, θα έχουμε ένα καινούριο πράγμα, ένα καινούριο πρόγραμμα με μεγαλύτερο πεδίο. Ε, θα αφορά όχι μονάχα την έρευνα αλλά και την καινοτομία και βεβαίως την ικανότητα Συγγνώμη, την οικοδόμηση ικανοτήτων. Αυτό είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό είναι πολύ ενδιαφέρον να στηρίξουμε, ε, και αυτό άλλωστε είναι ένας από τους κύριους στόχους μας, να στηρίξουμε συμμετέχοντες ε, που θα έχουν διαφορετικά επίπεδα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης ε, έχει ε, έχει αυξηθεί, έχει διπλασιαστεί η συμμετοχή των μη εθνικών ε, Ινστιτούτων Μετρολογίας, άλλων ε, Ινστιτούτων ή άλλων οργανισμών. Είπα και προηγουμένως ότι έχουμε πανεπιστήμια, έχουμε επιχειρήσεις, ήδη είναι περίπου χίλιοι συμμετέχοντες και ελπίζω ότι στο μέλλον θα αυξηθεί έχουμε διάφορα modules, διάφορα κομμάτια τα οποία αποτελούν το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Μετρολογίας. Ε, ε, το πρώτο μόντιουλ αφορά την επιστήμη. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα στο Πεκίνο ε, και είδα αυτά τα νέα εργαλεία μετρήματος με, το, με νερό επάνω και αστραγγίζεται το νερό και ανάλογα με το χρόνο που παίρνει για να αστραγγιστεί αλλάζει, μπορείς να κάνεις πιο σωστή μέτρηση. Έχουμε επίσης το δεύτερο μόντουλ που είναι η καινοτομία. Θέλουμε να κάνουμε κοινέ δράσεις με την βιομηχανία έτσι ώστε να μπορέσει η ευρωπαϊκή καινοτομία να βρει το δρόμο της. Όσον αφορά την τυποποίηση, το είπα και προηγουμένως, η Μετρολογία έχει συμφωνία με το Σένσεν και ελπίζουμε ότι σύντομα θα συνεργαστούμε και με το έτσι, έτσι ώστε να μπορέσουμε ε, να αναπτύξουμε και στρατηγική όσον αφορά την ε, ανταγωνιστικότητα της ε, καινοτομίας. Ε, το, επίσης ασχολούμαστε με την έρευνα πριν από τον καθορισμό ρυθμίσεων και τα λοιπά και το τελευταίο το οποίο μας απασχολεί είναι όπως είπα και προηγουμένως η οικοδόμηση ικανοτήτων. 30% των χρημάτων της ε, Κομισιόν θα ε, δαπανηθούν ε, για την συμμετοχή μη μετρολογικών Ινστιτούτων. Βεβαίως ένα μεγάλο κομμάτι των χρημάτων θα έπρεπε να πάει στην ε, διαχείριση, αλλά δεν θα το κάνουμε. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε το μεγαλύτερο κομμάτι των χρημάτων έτσι ώστε να συνεργαστούμε με εξωτερικούς συνεργάτες, με μετρολογικά ιστιτούτα Αυτά ήθελα να σας πω. Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες από αυτά τα λίγα που σας είπα τώρα, ε, μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μου, έχετε το email μου. Όμως, τελειώνοντας να πω ότι εδώ έχουμε μπροστά μας μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρόκληση γιατί ε, το δυναμικό που ανοίγεται μπροστά μας, που περιέχεται μάλλον σε αυτή ε, την ε, πρόταση είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι πρόκληση και μεγάλη ευκαιρία συνάμα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Ευχαριστώ που μου δώσατε την δυνατότητα να σας πω τα λίγα που σας είπα και εδώ οι συνάδελφοί μου μπορούν να πάρουν το λόγο να κάνουν κάποια επιπλέον σχόλια. Εγώ τελείωσα τα δικά μου σχόλια. Αυτή ήταν η παρουσίασή μου. Πρόεδρος. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε τον κύριο Χωσάινε για την παρουσίαση που μας έκανε. Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να πάρει το λόγο. Μπορούμε να ξεκινήσουμε την πρώτη συζήτηση. Θέλει κάποιος συνάδελφος να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ. Η διεθνής μετρολογία και η έρευνα υποτιμώνται αυτό φαίνεται ίσω και από το πόσοι παρόντε είναι μεταξύ των συναδέλφων μου. Πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε κάτι περισσότερο για να ενημερώσουμε την κοινή γνώμη. Δεν θυμάμαι πριν από πόσα χρόνια είχα την ευκαιρία να ασχοληθώ μαζί με τον Σάλφο Τσίτσεστερ με την οδηγία για τα όργανα μέτρησης. Είπαμε ακριβώς ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν τα ίδια επίπεδα σφάλματος για τα βενζινάδικα, για τις αντλίες τα βενζινάδικα, για το πόσο, πόση βενζίνη και μετά πόση βενζίνη αγοράζει κανείς. Και μετά από την ε, υπερψήφιση, δύο μέρες, ε, ε, διάβασα στην ε, ε, μια γερμανική εφημερίδα ότι η, η, η πετρελαιοβιομηχανία μαζί με τους ευρωβουλευτές θέλουν να κλέψουν τους καταναλωτές γιατί στη Γερμανία είχαμε λιγότερο ποσοστό σφάλματος κατά τη μέτρηση της ποσότητας βενζίνας που αγοράζει κανείς. Ξέρω ότι εδώ και 20 χρόνια έχουμε αλλάξει τους ε, αγωγούς και τους σωλήνες για την ε, υδροδότηση και συζητάμε ε, τώρα τη νέα οδηγία για το θέμα της υδροδότησης και είχε προταθεί να, εισάγεται, να εισάγονται στο νερό ε, οι όντα χαλκού για να βοηθούν και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενος που δεν έχουμε πλέον ε, ε μολύβδινους σωλήνες για την υδροδότηση και έχουμε χάλκινους σωλήνες οι οποίοι είναι πολύ πιο υγιείς. Με αυτά τα δύο παραδείγματα θέλω να σας δείξω τι ακριβώς κάνουμε και τι αποφεύγεται μέσω των αρνητικών παραδειγμάτων που σας έδωσα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που ε, ενισχύεται αυτό που έλεγα και εγώ. που μας βοηθάτε να ε, προβάλλουμε την εργασία μας ακόμη περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Ο Σάλφος ε, Έρτζογκ. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, Πρόεδρε, να ενημερώσετε τις πολιτικές ομάδες ότι πρέπει να είναι παρόντες οι συνάδελφοι στις συνεδριάσεις που διοργανώνουμε. Ξέρω, δεν φταίτε εσείς. Αλλά ξέρετε, πολύ συχνά ε, κατηγορούμε τους ευρωσκεπτικιστές ότι αμαυρώνουν την εικόνα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Αλλά και η παρουσία μας σήμερα δεν βοηθάει. Είναι απαράδεκτη. Να ευχαριστήσω τώρα τον κύριο Χωσάιν για την παρουσία του και για την προετοιμασία. Η παρουσίαση ήταν θαυμάσια, το έγγραφο μας υποβλήθηκε ήταν πολύ ε, κατατοπιστικό. Μία ερώτηση. Οι πολίτες μας ε, έχουν ε, πολλά εξαρτήματα τεχνολογικά και ε, έχουν τόσα εργαλεία επάνω τους που και οι ίδιοι έχουν γίνει ένα είδος εργαλείου μέτρησης. Έχουμε τόσα κινητά και άλλα τεχνολογικά, άλλες τεχνολογικές συσκευές επάνω μας, που έχουμε γίνει και εμείς ε, όργανα μέτρησης. Είστε μια οργάνωση που νομίζω την ε, εμπιστεύονται πολύ οι πολίτες. Οπότε η ερώτησή μου, πώς να συμμετέχουν οι πολίτες στις μετρήσεις. Μάλιστα με ακρίβεια. Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την ε, κοινωνική πρόκληση, πώς θα τη συμπεριλάβετε στην εργασία σας. Ίσως ε, πλατιάζω λίγο, αλλά πραγματικά με ενδιαφέρει πώς ε, οι πολίτες μας θα συμμετέχουν στην επιστημονική, ε, στο επιστημονικό γίγνεσθε μέσω συμμετοχής της μετρήσεις. Ξέρετε, εγώ είμαι εισηγήτρια ε, για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Συζητάμε λοιπόν για τη χρηματοδότηση της έρευνας. Θα ήθελα να τονίσω ότι το Κοινοβούλιο δεν θα υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό αν δεν δούμε δέσμευση από πλευράς του Συμβουλίου ότι θέλουν να υπάρξει σε προκαταρκτική φάση μεγάλη χρηματοδότηση όλων των ε, πιστώσεων που θα μας βοηθήσουν να βγούμε από την κρίση και η έρευνα οπωσδήποτε είναι κάτι τέτοιο. Παίζεται λοιπόν τέτοιο ρόλο ε, και ήθελα να είναι σαφές ότι θα σας βοηθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει και Πρόεδρος. Θέλουν άλλοι το λόγο. Όχι. Δεν υπάρχουν άλλοι. <laughs> Ε, Θεωρούμε ότι έκλεισε η συζήτηση. Θέλει κάποιος άλλος να πάρει το λόγο, θέλετε να δευτερολογήσετε. Ναι, να κάνω ένα σχόλιο. Ε, πραγματικά με απασχολεί ιδιαίτερα πώς να συμμετάσχουν οι πολίτες και οι πρότασή σας. Πώς θα συμμετάσχουν δεν μπορώ να σας απαντήσω, αλλά κάτι μπορεί να σε ενδιαφέρει είναι ότι είναι πολύ πιο εύκολο τα όργανα μέτρησης να είναι ε, άψυχα. Αν είναι έμψυχα είναι πιο δύσκολη η μέτρηση. Αλλά υπάρχει ένας κλάδος που λέγεται ήπιας μορφής μετρολογία ε, δεν είναι πράγματα τα οποία πιάνει κανείς. Για παράδειγμα πώς μετράμε τον πόνο. Σε ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προείδρευσα μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για να εκπονήσουμε ένα έγγραφο για τη μέτρηση του πόνου. Πώς ε, μετράτε το επίπεδο ε, ευημερίας, ε, συγγνώμη, όχι, το επίπεδο ε, Ευτυχία των ανθρώπων. Γιατί είναι σημαντικά αυτά τα θέματα. Υπάρχουν τομείς όπου μπορούμε να τα εξετάσουμε αυτά για να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη μεθόδων ε, μετρήσεων που να είναι διαφορετικές από τις μετρήσεις της φυσικής αλλά όπου θα συμμετέχουν οι πολίτες. Μπορούμε να το εξετάσουμε. Είναι κάτι που θα μπορούσαμε να εξετάσουμε. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε. Οπωσδήποτε. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Ευχαριστούμε τον ε, κύριο Καμάλο Σέιν, ο οποίος είναι πρόεδρος της ε, Euromet για την παρουσίαση που μας έκανε. Ολοκληρώσαμε λοιπόν αυτό το σημείο της ημερησίας διατάξεως, τον ευχαριστούμε και τον αποχαιρετούμε. Και περνάμε λοιπόν στο επόμενο σημείο. Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριο Χωσέ. Allora, passerei al rapporto di Ford. Θα περάσουμε τώρα στην έκθεση της συναδέλφου Βίκη Φόρντ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Um, Δεν έχουμε πάρα πολλούς παρόντες στην αίθουσα. Να ευχαριστήσω όσους είναι εδώ. Έχουμε κάποιες τροπολογίε. Ε, θα εκπονήσουμε για κάποιες συμβαστικές ε, τροπολογίε, Έγινε συζήτηση σήμερα το πρωί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Θα ήθελα ε, να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες που υπονοούν ότι δεν είναι ακριβές οι εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα. Σήμερα όμως οι δικοί μας είπαν πως εάν οι εταιρείες παραγωγής ενέργειας δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τεχνολογία αποθήκευσης και δέσμευσης του άνθρακα, αλλά πρέπει να βασιστούν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην πυρηνική ενέργεια όπου αυτό επιτρέπεται, τότε το κόστος των επενδύσεων για τις υποδομές ε, θα αυξηθεί κατά 40% βάσει των δικών τους εκτιμήσεων. Δεν λένε ότι όλες οι τεχνολογίες αποθήκευσης και δέσμευσης είναι φθηνότερες από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά κάποιες ε, τουλάχιστον και μπορεί να εκτιναχθεί το κόστος ε, Οπότε εγώ ε, θα αντιταχθώ στις τροπολογίες ε, που υπονοούν ότι είναι ακριβή αυτή η τεχνολογία γιατί δεν συνάδει αυτό με τη γνώμη των ειδικών. Επίσης, αυτό που με ανησυχεί είναι ε, ότι δεν πρέπει να υπονομεύσουμε τη δήλωσή μας, δηλαδή ότι πρέπει να έχουμε στόχους τεχνολογικά ουδέτερους, διότι είχαμε ένα συγκεκριμένο στόχο που υποχρεώνει τους ανθρώπους να επενδύουν σε μία τεχνολογία ε, παραγωγική μείωση των εκπομπών περιορίζοντας έτσι τις επενδύσεις όλες τις υπόλοιπες τεχνολογίες. Νομίζω ότι πρέπει να ε, είναι η χειρή δήλωση. Θα κάνουμε γι' αυτό ακριβώς το ζήτημα. Υπάρχουν και άλλες τροπολογίες που δεν κατανόησα πλήρως. Ε, Ε, για την ενθάρρυνση των βιομηχανιών που χρησιμοποιούν ε, τέτοιες ε, τεχνολογίες. Το ανθρακικό παραδείγματος χάρη, δεν υπάρχουν και τόσες πολλές, έχουμε ήδη πολλά αναψυκτικά και ο κλάδος αυτός δεν είναι και τόσο μεγάλος. Δεν είναι τόσο μεγάλο ε, το βάρος του κλάδου ώστε να πολλαπλασιαστούν τα προβλήματα. Δηλαδή ε, δεν πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας ε, στις βιομηχανίες που χρησιμοποιούν το ανθρακικό. Αντίθετα πρέπει να ασχοληθούμε στις τεχνολογίες αποθήκευσης και δέσμευσης για να μειώσουμε τις εκπομπές του διοξιδίου. Έχουμε ήδη συντάξει κάποιες συμβαστικές τροπολογίες, κάποιες θα χρειαστεί να τις ψηφίσουμε κυρίως τροπολογίες του σκιώδης ηγετή από τους ε, πράσινους ε, που ακολουθεί διαφορετική γραμμή ε, σε σχέση με τη γραμμή όλων των υπόλοιπων πολιτικών ομάδων. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Χέρτζοκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. συντομία, να πω ότι πρώτα μάλλον να ευχαριστήσω τη Βίκη για την έκθεση θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε συμβασμό για πολλά ζητήματα μέσα από τις συμβαστικές τροπολογίες. Θέλω να πω πως κάποιοι συνάδελφοι κατέθεσαν ε, τροπολογίες που κλείνουν από τη γραμμή των σοσιαλιστών, δηλαδή κατά των τεχνολογιών CCS, ενώ για αυτό το ζήτημα τουλάχιστον έχουμε θέση. Είμαστε υπέρ των τεχνολογιών αποθήκευσης και δέσμευσης ε, του άνθρακα. Θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα τμήμα της λύσης. Και αυτό που λείπει είναι να συνειδητοποιήσουμε πόσο επίγον είναι. Πρέπει να κινηθούμε ταχύτατα. Εγώ κατέθεσα ε, διάφορες τροπολογίες και μία συγκεκριμένα όπου λέω ότι σε κάποιες χώρες έχουν ληφθεί αποφάσεις για τα πυρηνικά ε, και έχουμε και το φθηνό σχιστολιθικό αέριο και χρησιμοποιούμε πολύ περισσότερο άνθρακα και αν ακολουθήσουμε αυτή την άγουσα είναι ακόμη πιο κατεπήγον το να ε, χρησιμοποιήσουμε αυτή την τεχνολογία CCS. Πρέπει να αποφασίσουμε. Αν θέλουμε να χρησιμοποιούμε περισσότερο άνθρακα, τότε χρειαζόμαστε το CCS. Ε, για την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα, δεν μπορεί να νουραγώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση υπό αυτό το πρίσμα θα ε, εξετάσουμε τις τροπολογίες και θα βρούμε επικοδομητικές λύσεις σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους και με την εισηγήτρια ώστε να ολοκληρώσουμε γρήγορα ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα στα κράτη-μέλη ότι οποιασδήποτε και αν είναι οι δημόσιες απόψεις που έχουν καθυστερήσει τα προγράμματα δεν μπορούμε να καθυστερούμε τη βιομηχανία, δεν μπορούμε να αμφισβητούμε το ότι είναι υψηλέ οι εκπομπέ ε, του διοξιδίου στη βιομηχανία. Είναι σημαντική η τεχνολογία δέσμευσης, ε, αποθήκευση και δέσμευση του άνθρακα. Ευχαριστώ κυρία Ερτζοκ Εάν δεν υπάρχουν ε, Α, θέλετε να πάρετε το λόγο πριν να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α, ο κύριος Βιδελ Κουάντρας, εντάξει, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν εξετάσουμε τις τροπολογίες, είναι σαφές ότι η δέσμευση και η αποθήκευση του άνθρακα δημιουργεί κάποιες διχογνωμίες ως τεχνολογία. Όλοι συμφωνούμε ότι η τεχνολογία αυτή ακόμη δεν έχει πλήρως αποδείξει ότι είναι η καλύτερη μέθοδος για να μειώσει τις εκπομπές μας με λογικό κόστος. Αλλά η αξιοποίηση αυτής της μεθόδου πρέπει να διερευνηθεί γιατί τα ορυκτά καύσιμα θα συνεχίσουν να είναι το μεγαλύτερο τμήμα του ενεργειακού μας μείγματος για τις επόμενες δεκαετίες. Είτε το θέλουμε είτε όχι συμμερίζομαι τις ανησυχίες που εξέφρασαν κάποια μέλη για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις αυτής της μεθόδου στις ε, τιμές της ενέργειας. Όμως οι τιμές αυτές ήδη επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό από τους φιλόδοξους στόχους μας για τη μείωση των ε, αερίων θερμοκηπίου και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Άρα πρέπει να βρούμε λύσεις. Όλες αυτές οι λύσεις προς το παρόν αυξάνουν το κόστος της ενέργειας. Επιπλέον, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας τονίζει ότι οι συμπληρωματικές επενδύσεις που χρειάζονται για την, ε, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για να ε, εμποδίσουμε την αύξηση κατά πάνω από δύο βαθμούς θα χρειαστεί να αυξηθούν περαιτέρω κατά 30% αν δεν έχουμε αυτή τη μέθοδο στη διάθεσή μας. Παρόλα αυτά η μέθοδος αυτή, για όλα αυτά μάλλον, ε, μάλλον. παρόλα αυτά, για να δούμε αν θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη μέθοδο, πρέπει να δούμε πόσο θα κοστίσει. Άρα, πρέπει όχι μόνο να αναπτύξουμε περαιτέρω αυτή την τεχνολογία για τη δέσμευση του διοξίδιου του άνθρακα, αλλά να εξετάσουμε και σε τι θα μπορούσε να χρησιμεύσει αυτό το αέριο όταν θα δεσμευθεί. Αυτό το αναφέρουν μερικές τροπολογίες. Συνολικά, κυρία Πρόεδρε. Δεν τα δίνουμε όλα για τη μέθοδο αυτή, αλλά να τις δώσουμε μια ευκαιρία. Ευχαριστώ. Πρώτα η Επιτροπή ή πρώτα η κυρία Φόρντ. Α, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ε, νομίζω ότι ακούσατε τις δύο μεγάλες ομάδες του Κοινοβουλίου. Βοηθάει λοιπόν και λένε ότι πρέπει να στηριχθεί αυτό. Υπάρχουν τροπολογίες από τους πράσινους που δεν είναι ιδιαίτερα υπέρ της ε, δέσμευσης και αποθήκευσης και μια τροπολογία επίση από πλευρά σοσιαλιστών που είναι κάπως ε, επίσης σκεπτική αλλά από ό,τι κατάλαβα την ε, εκπρόσωπό τους δεν είναι η άποψη της ομάδας. Οπότε περιμένω ότι η Επιτροπή μας θα δώσει ιδιαίτερα σαφές μήνυμα προς την Κομισιόν ότι θα θέλαμε επίγουσα δράση ιδιαίτερα για μερικά από τα ε, προγράμματα επίδειξης ε, της τεχνολογίας ε, αυτής. Και παρακαλώ, κύριοι της Επιτροπής, κύριε, κυρίες και κύριοι της Επιτροπής, καταλαβαίνω ότι περιορισμούς έχει η Κομισιόν όταν πρέπει με βάση χρονοδιαγράμματα να χορηγήσουν πιστώσεις. Αλλά η τεχνολογία αυτή έχει σοβαρά θέματα περίπλοκου προγραμματισμού. Είναι λοιπόν σημαντικό να σεβαστούμε τις διαδικασίες των κρατών μελών όταν λαμβάνουν αποφάσεις για τον προγραμματισμό της δράσης τους, ε, για μελέτες, για παράδειγμα, γεωλογικές σε διάφορες περιοχές. Αυτά τα θέματα είναι πολύ περίπλοκα για την ε, ε, δέσμευση του διοξίδου του άνθρακα παρά για πολύ πιο απλά προγράμματα και έχω την εντύπωση ότι οι προθεσμίες δεν μπορούν να τηρηθούν για διάφορα, μερικά, για διάφορα προγράμματα που συζητιούνται. Καταλαβαίνω ότι θέλετε να προχωρήσει το θέμα, αλλά είναι πολύ περίπλοκα τα προγράμματα και αυτό πρέπει να το σεβαστούμε. Πρέπει λοιπόν ως Κοινοβούλιο να υποστηρίξουμε λίγο περισσότερη ευελιξία για τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστούν οι ε, προθεσμίες. Γιατί αν οι προθεσμίες αυτές είναι ανέφικτες, δεν θα γίνει τίποτα τελικά. Γιατί αντιμετωπίζουμε γραφειοκρατικά τυπικά τα θέματα. Να εξετάσετε και αυτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ακού, άκουσα με προσοχή όλες τις απόψεις που εκφράστηκαν. Θα ήθελα εξ ονόματος της Επιτροπής να σας πω ότι αυτή η ανακοίνωση για την δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα ε, είχε, ξεκίνησε από την ε, αναγνώριση της ανάγκης να συζητηθεί το θέμα αυτό. Βεβαίως καλωσορίζουμε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γνωρίζοντας πάντως ότι αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να διαχειριστούμε τα υφιστάμενα προγράμματα πόρων και δραστηριοτήτων που έχουν ήδη ξεκινήσει δηλαδή, αλλά είναι και μια πάρα πολύ θεμελιώδης ε, στιγμή γιατί ε, ξεκινάει ο σχεδιασμός μελλοντικών δραστηριοτήτων, εκ των οποίων θα ήθελα να αναφέρω δύο-τρεις. Συζήτηση έγινε για το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο σε λίγο ολοκληρώνεται για τα έτη 2014 έως 2020 και επομένως με τον τρόπο αυτό θα έχουμε περισσότερες δυνατότητες στήριξης των σημαντικών νέων τεχνολογιών που θα μας οδηγήσουν προς μια ελεύθερη από διοξίδιο του άνθρακα ατμόσφαιρα πράγμα για το οποίο έχει δεσμευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το δεύτερο είναι ότι προσπαθούμε τώρα να καθορίσουμε ε, το πλαίσιο για το κλίμα που θα αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 2020-2030. Ε, το ρόλο που θα παίζουν τα ορυκτά καύσιμα, το ρόλο που θα παίξει η δέσμευση αποθήκευση άνθρακα, ε, ναι, καινοτόμες μορφές, ε, καινοτομίες μάλλον που θα αφορούν την ενέργεια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κτλ. Ίσως να προσθέσω και δύο-τρία άλλα πράγματα, γιατί άκουσα διάφορα ενδιαφέροντα, γράφει και ενδιαφέροντα η πρόταση εδώ. Υπάρχει σίγουρα ε, διάδραση ανάμεσα στην τεχνολογία, δέσμευση, αποθήκευση άνθρακα και τις ε, νέες μορφές, ε, ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Η Κομισιόν καταλαβαίνει ότι δεν θα πρέπει να δούμε τις τεχνολογίες αυτές σαν ανταγωνιστικές κατά την άποψή μα, ε, η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, οι τεχνολογίες που συνδέονται δηλαδή με το CCS και οι τεχνολογίες που συνδέονται με την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να ειδωθούν ως ε, ε, συμπληρωματικέ έτσι ώστε το ενεργειακό μείγμα να προκύψει με όσο γίνεται πιο καλό και αποτελεσματικό τρόπο. και ε, έχουμε και πολιτική στήριξη όσον αφορά την ενσωμάτωση αυτών των δύο δυνατοτήτων. Όσον αφορά τώρα την παρούσα κατάσταση των προγραμμάτων ε, και τα τελευταία σχόλια που είπε η κυρία Φόρτ σχετικά με την δυνατότητα μεγαλύτερης ευελιξίας και παροχή περισσότερων επιλογών γενικώ ομιλούντες ε, τα ενεργειακά προγράμματα σε όλες τις επιλογές τους είναι περίπλοκα. Υπάρχουν οι διαδικασίες αδειοδότησης ε, και ε, διάφορες διεργασίες οι οποίες είναι περίπλοκες και σε τοπικό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο των κρατών μελών δηλαδή. Το θέμα της δέσμευσης και αποθήκης του άνθρακα δεν αλλάζει, δεν είναι κάτι καινούριο. συζητιέται ήδη εδώ και αρκετό καιρό και ξέρουμε ότι έχουν υπάρξει σημαντικές αργοπορίες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα συνεχίσουμε ή ότι δεν προτιθέμεθα να συνεχίσουμε ή ότι δεν θα στηρίξουμε περαιτέρω τις προσπάθειες ε, οι πολιτικές οι οποίες ε, ήδη προετοιμάζονται τώρα προς αυτή την κατεύθυνση οδηγούν και θα υπάρξουν και νέες ε, δράσεις οι οποίες τώρα συζητιούνται. Ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρος. Κυρία Φόρτ, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Όχι. Άψογα. Να υπενθυμίσω λοιπόν ότι στις 5 Νοεμβρίου θα ψηφίσουμε στην ε, Επιτροπή. 5 Νοεμβρίου η ψηφοφορία. Και τώρα θα περάσουμε στο επόμενο θέμα μας. Α, ναι, η αποστολή στη Λιθουανία. Να πω λοιπόν στους συναδέλφους ότι μία αποστολή της Επιτροπής ε, Ήτρε, την οποία συμμετείχα και εγώ, μαζί με τη συνάδελφο Κολάσκα Μπομπίνσκα, τον κύριο Γκρίψε και τον συνάδελφο Ρόμπερτ Κοβάλε, ε, μια αντιπροσωπεία λοιπόν επισκέφθηκε το Βίλνιους από τις 15 μέχρι τις 17 Ιουλίου του 2013. Μεταξύ άλλων είχαμε και τους Μπασίλτης ε, και σε τους Λιθουανούς συναδέλφους. Συναντήσαμε στη διάρκεια της επίσκεψής μας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της ε, Λιθουανίας ο οποίος μας ακοινοποίησε το πρόγραμμα της Λιθουανικής Προεδρίας. Συναντήσαμε επίσης ε, διάφορους υπουργούς, τον ε, ε, Υφυπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, τον Υπουργό Οικονομικών, καθώς επίσης και εκπροσώπους οργανώσεων κλαδικών και τομεακών. Είχαμε κοινή συνεδρίαση με τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών της Επιτροπής Επιστήμης, ε, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού του Λιθουανικού Κοινοβουλίου. Επίσης συναντήσαμε τον Υπουργό Ενέργειας και τον Υπουργό Εκπαίδευσης και Επιστήμης. Ε, μέσω της επίσκεψης στο Βίλνιους, ε, τα μέλη που συμμετείχαν είχαν τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσουν τις ε, προτεραιότητες της Λιθουανίας σε τομείς που άπτονται των θεμάτων της Επιτροπής Ήτρα καθώς επίσης και να δουν σε βάθος την παρούσα κατάσταση στη Λιθουανία, καθώς επίσης και τις προκλήσεις της Λιθουανίας. Οι Επίσης, κατά τη διάρκεια της επισκέψεως, μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν στην ε, ενιαία αγορά ενέργειας, την πυρηνική ασφάλεια, την ασφάλεια της ε, ε, τροφοδοσίας ενέργειας, τα πολιετή προγράμματα και τα λοιπά. Θέλετε να προσθέσετε κάτι σε αυτά που ε, είπα ήδη για τη Λιθουανία. Όχι. Πάρα πολύ ωραία. Ε, ολοκλήρωσε λοιπόν η Επιτροπή της Εργασίας της. Σταματούμε λοιπόν για να ξαναρχίσουμε στις 5 με τους συντονιστές. Αύριο το πρωί ε, θα αρχίσουμε πάλι σαν ολομέλεια της Επιτροπής Ήτρε στις 9 σε κοινή και το απόγευμα θα έχουμε κοινή συνεδρίαση με την ΕΜΒΗ.